ευχαριστώ. Ξεκινάμε την ε, Ολομέλεια του Κοινοβουλίου που σταματήσαμε στις 5 Οκτωβρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες ε, της σημερινής Ολομέλειας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα θύματα των πυρκαγιών στα